Good morning. Uh, uh, Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Καλώς όρισαν οι συνάδελφοι των Επιτροπών ε, Πολιτικών Ελευθεριών και Δικαιωμάτων των Γυναικών για αυτή την κοινή ακρόαση. Με μεγάλη μας χαρά θα συμπροεδρεύσουμε με τον κύριο Μωράες και η συνεργασία των δύο επιτροπών μας είναι πάρα πολύ αγαστή. Για πολλά θέματα έχουμε συνεργαστεί και σήμερα πρόκειται να ασχοληθούμε με ένα θέμα από τα πιο σημαντικά κοινού ενδιαφέροντος η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ε, Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Βρισκόμαστε σε μια κομβική συγκυρία γιατί μετά την υπογραφή αυτής της σύμβασης τον Ιούνιο του 2017. Τώρα θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία στο Συμβούλιο και ένας κώδικας διοντολογίας όσον αφορά τους εφαρμοστικούς κανόνες αυτής της ε, σύμβασης από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να δούμε τι αποφάσεις θα ληφθούν στη συνέχεια για την ε, κύρωση της συνθήκης αυτής πάντως εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θέλουμε να μείνουμε σταυρωμένα τα χέρια. Θέλουμε να προκαλέσουμε μια πλήρη και σύντομη κύρωση της συνθήκης. Οπότε έχουμε την σημερινή παρουσίαση ε, από την νομική υπηρεσία. Θα είναι για τον σκοπό μας αυτό κάτι το πάρα πολύ σύντομο και τώρα να δώσω στον συμπρόεδρο τον λόγο. Μωράς, σε ευχαριστώ. Συνάδελφε, σήμερα με τους συναδέλφους των Επιτροπών θα ακούσουμε αυτή την παρουσίαση της νομικής υπηρεσίας. Θα υπάρξουν διευκρινήσεις όσον αφορά σημαντικές πτυχές της ε, εφαρμογή της συνθήκης Κωνσταντινούπολης. Στο ότι δηλαδή θα πρέπει συνολικά να προσχωρήσει σε αυτή τη συνθήκη, σε αυτή τη σύμβαση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να ακούσουμε επίση μια ανάλυση για τι αρμοδιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των κρατών μελών στην άλλη όσον αφορά το περιεχόμενο τη σύμβαση. Επίση, σα υπενθυμίζω, στι 4 Μαρτίου παρουσίασε δύο προτάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τη σύμβαση για την πρόληψη και καταπολέμηση βίσκα των γυναικών και οικιακή βία. Υπήρχε μια απόφαση του Συμβουλίου όσον αφορά την υπογραφή της σύμβασης και η άλλη επίση φορούσε την σύμβαση. Έχουμε τώρα στις 12 του 17 ένα ψήφισμα του Κοινοβουλίου όσον αφορά μια σειρά συστάσεων προς ε, Συμβούλιο, Επιτροπή και Κρατημέλη για λαμβάνεται υπόψη ότι η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόκειται να εξασφαλίσει ένα νομικό πλαίσιο συνεπές ώστε να υπάρξει πρόληψη και η καταπολεμιστή των γυναικών και της βίας κατά των γυναικών και της υποστήριξης των ε, θυμάτων ε, και την πλαισίωση από τις ε, εσωτερικές και εξωτερική πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τώρα να δώσουμε τον λόγο στην νομική υπηρεσία. Έχετε 12-15 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρίε και κύριοι. Η νομική υπηρεσία έλαβε μια, ένα αίτημα να εκδώσει νομ, ε, γνωμοδότηση από τους πρόεδρους των Επιτροπών ΛΥΠΕ σχετικά με θέματα που σχετίζονται με την υπογραφή της ε, σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, είναι μια σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης που έχει σχέση με την πρόληψη και την καταπολέμηση βίας κατά των γυναικών και της οικιακής βίας. Η σύμβαση έχει τεθεί σε εφαρμογή από τον Αύγουστο του 2014. Μέχρι τώρα όλα τα κρατημέλη Τις Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν υπογράψει τη σύμβαση, αλλά δεν την έχουν όλα επικυρώσει. Η σύμβαση είναι επίσης ανοιχτή, προκειμένου να υπογραφεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 75.1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολη στις 13 Ιουνίου 2017, επί τη βάση δύο αποφάσεων του Συμβουλίου. Στην Κορεπέρ, συνάντηση Κορεπέρ τον Απρίλιο του 2017, εκφράστηκαν διάφορες ανησυχίες για αυτές τις αποφάσεις του Συμβουλίου από την Κομισιόν. Η Κομισιόν αμφισβητεί την προσέγγιση που αφορά τι νομική, τις νομικές βάσεις την άσκηση των αρμοδιοτήτων από πλευρά Ευρωπαϊκής Ένωσης και το γεγονός ότι το Συμβούλιο είχε χωρίσει την απόφαση που αφορά την υπογραφή της σύμβασης σε δύο μέρη. Αυτό σημαίνει ότι το Συμβούλιο υιοθέτησε δύο διαφορετικές αποφάσεις. Μία που αφορούσε τα στοιχεία της σύμβασης σε ό,τι αφορά την δικαστική συνεργασία επί ποινικών θεμάτων και μία άλλη που αφορά τα θέματα ασύλου και μία επαναπρόθεσης. Η, το αίτημα γνωμοδότησης από πλευράς νομικής υπηρεσία καλύπτει ουσιαστικά παρόμοιες ανησυχίες. Σε αυτή την σύντομη παρουσίαση θα σας ε, ε, ε, δώσουμε με λησελίες γραμμές τα πορίσματά μας. Η πρώτη, αφορά, η πρώτη ερώτηση αφορά την σωστή ουσιαστική νομική τις σωστές ουσιαστικές νομικές βάσεις των αποφάσεων για την υπογραφή. Ε, θα θέλω να σας υπενθυμίσουμε ότι η σύμβαση της ε, Κωνσταντινούπολης είναι μια σφαιρική ε, ε, σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μεταξύ άλλων σχετίζεται με την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών, την προστασία και τη στήριξη των θυμάτων και επίσης τους ορισμούς των σχετικών ποινικών αδικημάτων. Επίσης υφίστανται στη Σύμβαση ξεχωριστά κεφάλαια για δικονομικό, με δικονομικές διατάξεις ε, και για τις μετανάστευση και το άσυλο. Επίσης συμπεριλαμβάνει θεσμικές διατάξεις ε, για, και έναν μηχανισμό παρακολούθησης. Η Κομισιόν λοιπόν πρότεινε η Σύμβαση να υπογραφεί επί τη βάση των άρθρων 82 παραφρος 2 και 84 Αυτές οι διατάξεις έχουν, σχετίζονται αντίστοιχα με τα δικαιώματα των θυμάτων ε, και το έγκλημα και την, πρόληψή του. Το Συμβούλιο όμως ε, έλαβε διαφορετική προσέγγιση ε, βάσισε την πρώτη απόφαση στο άρθρο 83 παράγραφος 1, δηλαδή μια νομική βάση που σχετίζεται με το ουσιαστικό ποινικό δίκαιο και το άρθρο 82 παράγραφος 2 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η λογική πίσω από την προσέγγιση αυτή του Συμβουλίου ήταν ότι εντόπισε τομείς που καλύπτονται από δύο οδηγίες ποινικού δικαίου ω ε, τομεί αποκλειστική αρμοδιότητα Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτέ οι οδηγίε αφορούν ε, το λαθρεμπόριο ανθρώπων και την σεξουαλική εκμετάλλευση. Το Συμβούλιο ε, εντόπισε αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο στο μέτρο που αυτά τα δύο κείμενα ε, αλληλεπικαλύπτονται, τις δύο οδηγίες αλληλεπικαλύπτονται με διατάξεις τη σύμβαση. Η δεύτερη απόφαση βασίστηκε στο άρθρο 78 παράγραφος 2 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Αυτές οι διαφορές μεταξύ των αποφάσεων που αλήθηκαν και οι διαφορετικές νομικές βάσεις εξηγούνται από τις διαφορετικούς, τους διαφορετικούς συσχετισμούς ψήφων στο Συμβούλιο εξαιτία τη ειδική θέση τη Ιρλανδία και του Βασιλείου. Αναλύοντα το θέμα των νομικών βάσεων, η νομική υπηρεσία βασίστηκε στην νομολογία του Δικαστηρίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Από αυτή την ανάλυση θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι η επιλογή τη νομική βάση πρέπει πάντοτε να βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρμόδια να υιοθετήσει μια συγκεκριμένη νομική πράξη, θα πρέπει να βασίζεται κατά κανόνα σε μία και μοναδική νομική βάση. Αυτή η νομική βάση θα πρέπει να είναι αυτή την οποία απαιτεί ο βασικός στόχος ή το βασικό στοιχείο της πράξης. Ε, κατ' εξαίρεση, αν αυτή η νομική πράξη ταυτόχρονα επιδιώκει αριθμό στόχων που συνδέονται με τρόπο που είναι αδύνατον να διαχωριστούν και με τρόπο όπου κανένας από αυτούς τους στόχους δεν είναι δευτερεύον έναν των υπολείπων, τότε ε, αυτή η νομοθετική πράξη πρέπει να βασίζεται στις αντίστοιχες νομικές βάσεις. Αυτό όμως είναι η εξαίρεση. Με άλλα λόγια, σύμφωνα με το δικαστήριο, πρέπει να εντοπιστεί το κέντρο βάρους της πράξης και αυτό θα αποφασίσει τη νομική βάση. Σύμφωνα με αυτή τη λογική, η νομική υπηρεσία διέτρεξε την σύμβαση και εντόπισε δύο βασικά δεσπόζοντα στοιχεία. Τα δικαιώματα των ε, ε, θυμάτων και δεύτερον το έγκλημα και η πρόληψή του. Αυτά είναι τα δύο βασικά στοιχεία, συστατικά στοιχεία της σήμασης από την πλευρά της υπογραφής και ε, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διατάξη για το άσυλο ε, είναι δευτερεύουσες κατά την άποψή μου. μας. Οι διατάξεις αυτές δεν είναι κυριαρχές στα στοιχεία της σύμβασης. Είναι, ε, σχετίζονται με ε, συντονισμό των πολιτικών και ολιστική απάντηση ε, και εμπίπτουν περισσότερο στο γενικότερο στόχο του σχεδιασμού ενός συνολικού πλαισίου πολιτικών και μέτρων για την προστασία και την συνδρομή σε όλα τα θύματα της βίας εναντίον των γυναικών και της οικιακής βίας. Επιπλέον, σε ό,τι αφορά το θέμα της ε, σχέσης μεταξύ των πρωτοκόλων ε, opt-out και την επιλογή της νομικής βάσης, το δικαστήριο έχει αναφέρει ότι το πρωτόκολλο υπαριθμών 21 για τη θέση του Ηνωμένου Βασίλειου και της Ιρλανδίας σχετικά με, την, με το χώρο ε, ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης δεν είναι εφαρμοστή δεν είναι δυνατόν να έχει οποιοδήποτε αποτέλεσμα στο θέμα της, ε, επί του θέματος της ε, ορθής νομικής βάσης για την υιοθέτηση της ε, επιμαχής απόφασης. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η νομική βάση ενός μέτρου, δηλαδή το κατά πόσον αυτή σχετίζεται ή όχι, αυτό που πρέπει να αξιολογηθεί επί τη βάση αντικειμενικών παραγόντων όπως ο βασικός ή κυρίαρχος στόχος του μέτρου και αυτή θα αποφασίσει το πρωτόκολλο και όχι το αντίστροφο. Οπότε δεν θεωρούμε ότι χρειάζεται χωριστή νομική βάση για το άσυλο. Σε ό,τι αφορά το, τις ε, διατάξεις ουσιαστικού ποινικού δικαίου, οι αποφάσεις για την ε, ε, υπογραφή της σύμβασης εντοπίζουν αποκλειστικές αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τομείς που καλύπτουν από δύο οδηγίες, όπως είπαμε. Όμως, το δικαστήριο έχει καταστήσει σαφές ότι η νομική βάση εσωτερικής νομοθεσίας καθορίζεται από το βασικό συστατικό τους. Ε, ενώ ο κανόνας που μπορεί πιθανώς να επηρεαστεί ε, μπορεί να είναι απλώς ε, δευτερεύον συστατικός από τη νομοθεσία. Όπως θα δούμε αργότερα, αναλύοντας τις ε, ευρωπαϊκές αρμοδιότητες. Τα κράτη-μέλη διατηρούν τις αρμοδιότητες τους αναφορικά με τις διατάξεις του ουσιαστικού ποινικού δικαίου της σύμβασης. Οι ελάχιστες εξαιρέσεις, δηλαδή ε, τα, αυτά που καλύπτονται από τις ε, δύο ανωτέρω οδηγίες, είναι δευτερεύοντα στοιχεία. Υπό το φω των ανωτέρων και σύμφωνα με το νομολογία του δικαστηρίου, ε, η προσθήκη του άρθρου 83 παράγραφος 1 ως ξεχωριστή νομική βάση για την υπογραφή τη σύμβαση δεν φαίνεται να είναι απαραίτητη από νομικής πλευράς. Συνοψίζοντα τα απορίσματά μα σχετικά με τις νομικές βάσεις έχουν ως εξής. Το άρθρο 82 παράγραφος 2 τη Συνθήκη Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τα δικαιώματα των θυμάτων, το έγκλημα και ενδεχομένω. Ε, δικαι... συγγνώμη, θυμάτων του εγκλήματο και ενδεχομένω το άρθρο 84 για την πρόληψη του εγκλήματο φαίνεται ότι είναι οι σωστοί νομικοί, οι σωστέ νομικέ βάσει για την απόφαση υπογραφή τη Σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη, όπω ακριβώ το πρότεινε η Κομισιόν. Τώρα, θέλω να δώσω το λόγο στον συνάδελφό μου για τα παρακάτω. Thank you very much. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Να συνεχίσω με το δεύτερο ερώτημά σας που θέσατε της εξωτερικής δηλαδή αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτα να τονίσω ότι η σύμβαση είναι μεικτή συμφωνία. Ένωση και χώρες μέλη έχουν και οι δύο αρμοδιότητες στο πεδίο εφαρμογή της ε, σύμβασης και σε μεικτές συμφωνίες συμβαλόμενα μέρη είναι και η Ένωση και οι χώρες. Το δικαστήριο δήλωσε ότι για τις υποχρεώσεις από τέτοιου του συμφωνίες οι χώρες μέλη πληρούν εντός του Ευρωπαϊκού Δικαιικού Συστήματος υποχρεώσεις που έχουν σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και η οποία έχει αναλάβει την ευθύνη για την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας. Επομένως, σύμφωνα με τις υποχρώσεις του, της Ευρωπαϊκής Συνθήκης και όχι του Διεθνούς Δικαίου, όσο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρμοδιότητα για να συνάψει τη σχετική σύμβαση. Και το λόγο αυτό, το ζήτημα της αρμοδιότητας που θέσατε είναι πολύ ενδιαφέρον. Όπως βλέπετε από την ανάλυση μας, το ζήτημα των εξωτερικών αρμοδιοτήτων σε μεικτές συμφωνίες είναι περίπλοκο. Στη νομική βιβλιογραφία αναφέρονται στην αποθέωση της περιπλοκότητας. Για τους σκοπούς της παρούσης λοιπόν θα περιοριστούμε σε μια σύνοψη των βασικότερων συμπερασμάτων μας. Εξάλλου, τονίζω ότι οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν φτιάξει έναν λεπτομερή χάρτη των ε, διατάξεων της ε, Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης που δίνει και μια πλήρη ανάλυση των αρμοδιοτήτων, αλλά δεν χρειάζεται περισσότερη. Ε, θα εξετάσουμε πρώτα λοιπόν τις, ε, τους περιοχές αποκλειστικής εξωτερικής αρμοδιότητας. Διότι όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποκλειστική εξωτερική αρμοδιότητα, οι χώρες μέλη δεν μπορούν να ε, συμμετέχουν σε, να αναλαμβάνουν μάλλον διεθνείς υποχρεώσεις. Στη βάση της ανάλυσης αυτής, το κεφάλαιο 4 και διάφορες διατάξεις του, άρθρου, κεφαλαίου μάλλον 6, έρευνα, ε, δίωξη, διαδικαστική ε, ε, ε, διοικονομική διατάξεις κτλ. εμπίπτουν στην αποκλειστική εξωτερική αρμοδιότητα της Ένωσης. Το ίδιο για αιτήσει ασύλου. Από την άλλη μεριά, οι χώρε μέλη φαίνεται να είναι ευρέω αρμόδιες για το κεφάλαιο 5 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης για το ουσιαστικό ποινικό δίκαιο. Η οποία Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης περιλαμβάνει και το κεφάλαιο 9 που επιγράφεται monitoring mechanism. Το κεφάλαιο αυτό προβλέπει ομάδα εμπειρογνωμόνων για την δράση κατά της βίας κατά των γυναικών, που λέγεται Γκρέβιο, και επίσης Επιτροπή των Συμβαλωμένων Μερών που θα συντίθεται από προσώπους τους. Σε ό,τι αφορά τέτοιες διατάξεις, το δικαστήριο έχει καταστήσει σαφές ότι οι διατάξεις αυτές είναι επικουρικού χαρακτήρα και για το λόγο αυτό εμπίπτουν στην ίδια αρμοδιότητα όπως οι ουσιαστικές διατάξεις, ουσιαστικού δικαίου δηλαδή. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρμοδιότητα να προωθεί και να στηρίζει τις δράσεις των χωρών μελών στο πεδίο της πρόληψης του εγκλήματος, αποκλείοντας ωστόσο οποιαδήποτε εναρμόνιση. Τρίτη ερώτηση. Σχετικά με τους ενδεχόμενους νομικούς λόγους για την υιοθέτηση δύο διαφορετικών αποφάσεων για την υπογραφή της συμβάσεως. Όπως εξηγήσαμε προηγουμένως, η ειδική κατάσταση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας φαίνεται πως είναι ο λόγος, για τη διάσπαση της προτάσεως της Κομισιόν. Χωρίς να πω σε λεπτομέρειες, τονίζω ότι η προσέγγιση αυτή δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται από την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Και η διάσπαση αυτή, επομένως, δεν είναι αναγκαία από νομική άποψη. Μία απόφαση στην βάση του άρθρου 82, παράγραφος 2 τη συνθήκη τη Ένωση και ενδεχομένω και το 84 θα αρκούσαν Τέλος, η τέταρτη ερώτηση μας ζητεί να αναλύσουμε τις διαφορές μεταξύ της, Ευρωπαϊκής, δηλαδή της, Ευρω... της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και σε άλλο νομοθέτημα, δηλαδή τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των προσώπων με αναπηρίες. Εδώ υπάρχουν κάποιες βασικές διαφορές και θα ολοκληρώσω την παρουσίασή μου με την ε, απαρίθμηση αυτών των διαφορών. Πρώτο, σε ό,τι αφορά την ε, Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών η κοινή άσκηση ε, αρμοδιοτήτων στον χώρο που προβλέπεται για την Σύμβαση των, ε, της Κωνσταντινούπολης. Εκεί οι χώρες μέλη διατηρούν πλήρως τις αρμοδιότητες της εκτός του χώρου της αποκλειστικής αρμοδιότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις αποφάσεις για την υπογραφή της Σύμβασης Κωνσταντινούπολης. Δεύτερο, σε ό,τι αφορά τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταθέσει δήλωση αρμοδιοτήτων και έχει εγκρίνει δεοντολογικό κώδικα σχετικά με τι ρυθμίσει για τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χωρών μελών. Οι αποφάσει του Συμβουλίου για την υπογραφή τη Σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη δεν παραπέμπουν σε τέτοια έγγραφα. Α σημειωθεί ωστόσο ότι ενώ η δήλωση αυτή δεν απαιτείται από την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ωστόσο όπου αυτό είναι αναγκαίο, αποτελεί μια χρήσιμη βάση παραπομπής. και στις συμφωνίες που έχουν σχέση με δήλωση αρμοδιότητας ένωσης βρίσκουμε συνολικά καμιά εκατοστή τέτοιες. Άρα είναι μια πρακτική η οποία έχει πλέον ε, ε, κυρωθεί. Τέλος, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προβάλει επιφυλάξεις για την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, δεν αναφέρονται οποιασδήποτε σχετικές επιφυλάξεις στις αποφάσεις του Συμβουλίου για την υπογραφή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Εδώ ολοκληρώνουμε την παρουσίαση των βασικών συμπερασμάτων της νομικής μας έρευνας. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας και είμαστε στη διάθεσή σας για να φωτίσουμε περισσότερες λεπτομέρειες και να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Η πρόεδρος της Επιτροπής Γυναικών, ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας και τώρα πριν ε, δώσουμε το λόγο στα μέλη θα πρέπει να δώσουμε το λόγο στους συνεισηγητές για τη σχετική έκθεση που αφορά την σύμβαση του Ξέντινου Πόλεως. Κυρία Κορατσαβίλη, κυρία Μποναφόρε. Πρώτα πρώτα η κυρία Μπονφά. Έχετε τελευταία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι, σας ευχαριστούμε για την τόσο πλήρη σας ε, παρουσίαση. Τον Ιούνιο του 2017, αντί ε, για ένα, έφτιαξε δύο έγγραφα το Συμβούλιο, γιατί αυτό το θέμα το σημαντικό αφορά εκατομμύρια γυναίκες και ε, με την Κόρα Τσαμπίλ και τους και οδησυγητές ε, είχαμε κάποιε επιφυλάξει για αυτά τα δύο έγγραφα και όχι μόνο εμείς γιατί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απείλησε με αίτηση διευκρινήσεων από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το οποίο δεν έγινε. Οπότε τώρα έχουμε την δική σα νομοδότηση αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι πέρασε ένας χρόνος από τότε που ζητήθηκε αυτή η γνωμοδότηση και ακόμα παραμένει επίκαιρη για το θέμα δεν έχει ρυθμιστεί. Και αν επομένω εμεί επιμένουμε που το κάνουμε, γιατί ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ε, την κατονομή των αρμοδιοτήτων γιατί θα πρέπει να δούμε συγκεκριμένα πώς θα ισχύσουν τα της ε, Συμβάσκου για τις γυναίκες και θα πρέπει επίσης να παρακολουθήσουμε το αν υπάρχει πρόοδος ή αν υπάρχει πίσω γύρισμα. Τώρα, τι μάθαμε σήμερα, ότι αυτέ μας οι εμβολίε είναι βάσιμε και είχαμε μεγάλη πλειοψηφία όταν ε, εγκρίθηκε σχετική έκθεση και δεν υπάρχει κανένα λόγο να μην προχωρήσουμε έτσι και το Συμβούλιο αυτό το οποίο τα έκανε χωρίς να τα δικαιολογήσει και έτσι αδυνατίζει η θέση μας και αδυνατίζει και το κύρος της ε, συμβάσεως. Χρειάζεται μια συνολική προσέγγιση γιατί ε, αφορά όλες τις εκδηλώσεις στην βιομηχανία, την κοινωνία, τόσο ώστε να καταπολεμηθεί η βία κατά των γυναικών. Οπότε ε, η σύμβαση αυτή είναι ένα βήμα πρόοδου, αλλά θα πρέπει να υπάρξει στην πράξη βοήθεια. Με την ευκαιρία αυτή θα πρέπει να πούμε στα κράτη-μέλη τα σχετικά, γιατί ε, ήδη απευθυνθήκαμε στην Βουλγαρική Προεδρία με την σύνηση για να τους ε, πούμε ότι ανησυχούμε και εμείς όπως και η Επιτροπή δεν πήραμε απάντηση. Ε, νομίζω ότι τα νομικά θέματα είναι μια πρόφαση και ε, έτσι δεν γίνεται να υπάρξει και συνθήκε από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, τα πράγματα έχουν παγώσει για ένα νομικιστικό θέμα. Και κρύβεται πίσω από αυτό το Συμβούλιο και έτσι ε, μπλοκάρει για λόγους πολιτικούς την πρόοδο. Η αλήθεια είναι ότι η καταπολέμηση της βίας των ενεργών δεν είναι για τα κρατημέλη μια ε, προτεραιότητα. Και ακόμα χειρότερα, ανοιχτά λένε ότι δεν θέλουν να ακυρώσουν γιατί υπάρχουν κρυφοί ιδεολογική λόγια και υπενθυμίζω ότι και η βουλγαρική ε, ε, κυβέρνηση που τώρα που έχει την Προεδρία δεν πρόθεσε το σχετικό νομοσχέδιο. Να, γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και με, με τους συνεισυχητές στείλαμε την επιστολή στη Βουλγαρία, δεν πήραμε απάντηση και επίσης ο αρμόδιος επίτροπος και αντιπρόσωπος του ε, Δικαστηρίου της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μας μίλησε εδώ με ενθουσιασμό ευτυχώς αλλά στην ε, Κροατία παρά τις διαδηλώσεις τους δρόμους ε, και όσοι γίνονταν οι διαδηλώσεις κύρωσε την συνθήκη. Όταν λέμε για το φίλο δεν κρύβεται τίποτα πίσω από αυτό. Το κάνουμε για αυτή την ε, βία που στέφτηκα των γυναικών, που δυσανάλογα της ε, πλήση ως φαινόμενο. Δεν ε, θέλουμε να καταπολεμήσουμε την παραδοσιακή οικογένεια, αλλά την απειλή της βίας. Και στις 18 Μαΐου θα έχουμε την πρώτη επέτειο της προσυπογραφής ε, τη Συμβάση του πόλη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζω ότι μέχρι τότε θα έχουμε αποσπάσει κάποια αποτελέσματα και θα έχουμε πάρει την κατεύθυνση τη ε, κύρωσης και ελπίζω ότι τα κράτη-μέλη θα ακούσουν αυτό το οποίο λέμε σήμερα. Thank you very much, Mr. Ε, ευχαριστώ κυρία Συμπρόεδρε, συμφωνώ 100% με όλη μου την καρδιά όλα τα οποία ακούσαμε από την Κριστίν, την συνεισήγητρα. Ευχαριστούμε και την νομική υπηρεσία. Επιβεβαίωσε τις επιφυλάξεις μας, τις αμφιβολίες μας, τεκμηριωμένα, με επιχειρήματα νομικά, σε σχέση με το ότι τόσους δεσμούς υπάρχει από τα κατημέρια για την προσυμπογραφή και για την κύρωση της σύμβασης. Το θέμα είναι ότι η προσβογραφία δεν είναι τελική φάση αυτής της διαδρομή. Θα πρέπει να γίνει η κύρωση για να ολοκληρωθεί η προσχώρηση στην ε, σύμβαση. Οπότε είναι θέμα διαπραγμάτευσης με το Συμβούλιο. Και ακριβώς όπως είπε και η Κριστίν, δεν μας έχουν απαντήσει. Απευθύνω έκκληση στους συμπροέδρους μας. Εάν συμφωνείτε επί τη βάση της ε, γνωγότης νομικής υπηρεσίας και μια που με τόση πλειοψηφία το Κοινοβούλιο ενέκρινε το σχετικό κείμενο τον ε, Σεπτέμβριο, να απευθυνθούμε στον Πρόεδρο Ταγιάννη, στην Βουλγαρική Προεδρία, να ζητήσουμε, να τεθεί επί της τραπέζης, να συζητηθεί στο Συμβούλιο, να μπει στο θεματολόγιο του Συμβουλίου, μέσα διάταξη να επιταχυνθεί η πρόοδος προς, μια, προς ένα κώδικα διοντολογίας. Ήταν ιστορικά αυτά τα οποία έχουν γίνει, όπως είπε και η Κριστίν, γιατί φορούσε όλες τις γυναίκες και τις ανηλικές γυναίκες, όλους που έχουν πέσει θύματα αυτής από τρόπες βίας. Είναι απαράδεκτο να έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος και να έχουν γίνει τόσα λίγα. Σας υπενθυμίζω ότι μιλώ για γυναίκες οι οποίες σκοτώνονται, ε, ακροτηριάζονται, βιάζονται, ξαναγκάζονται σε γάμους, παρενοχλούνται, δένονται ε, και δεν μιλούμε για κάτι ιδεολογικό ή θρησκευτικό. Είναι σημαντική σημασία γιατί είναι το μόνο εργαλείο του διεθνούς δικαίου για αυτό το φαινόμενο. Έχει συγκεκριμένα μέτρα για το πώς ε, θα υπάρξει πρόληψη και προστασία καταπολέμηση της ετοιμορρησίας. Κανένα κρατός μέλος δεν κάνει αρκετά προς αυτή την κατεύθυνση. Κύπρος, Γερμανία, Κροατία προχώρησαν και άρα με, με πυγμή προωθήθηκε στην Κροατία το θέμα και όμως έχουμε πολλά κράτη-μέλη τα οποία δεν προχώρησαν προς την ακύρωση. Άρα Επαναλαμβάνουμε για το θέμα της βίας και των γυναικών. Δεν πρέπει να παρερμηνεύεται η σύμβαση. Πριν την ευκαιρία της επαιτίου της 8 Μαρτίου, ο πρόεδρος Ταγιάννη μίλησε στο Κοινοβούλιο και κάλεσε τον διαμεσολαβητή, το, το Συμβουλίο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι οποίοι τελικά ε, διευκολύνουν διευκρίνησαν το ότι όταν μιλούμε για φίλο δεν υποκρύπτεται κάτι άλλο. Απλώς εδώ προσπαθούμε να προστατεύσουμε αυτά τα οποία είναι σωστά να περιβάλλουν τις γυναίκες γιατί ο σοβινισμός είναι κάτι το οποίο απειλεί τις γυναίκες και όχι τις ε, οικογένειες. Άρα είναι σημαντικό να μείνουμε συσπηρωμένοι, ενωμένοι στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρχίσουν έναν δημιουργικό διάλογο, να καμφθούν οι σχετικές αντιστάσεις και ε, κάποιων ομάδων θρησκευτικών γιατί όπως είπε η Κριστίν είναι απαράδεκτο το ότι η Προεδρία του Συμβουλίου έχει παγώσει το θέμα της διαδικασίας κύρωσης. Και ολοκληρώνω λέγοντα ότι και η Κριστίν και εγώ μένουμε προσιλωμένοι σε αυτόν τον σκοπό, αλλά και άλλοι εδώ. Θέλουμε να υπάρχει μηδενική ανοχή όσον αφορά τη βία των γυναικών. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κοράτσα Βίλτ, θα εξάγουμε τα κατάλληλα συμπεράσματα. Θα ήθελα να ρωτήσω τα, τα άλλα μέλη αν θέλουν να λάβουν το λόγο μετά από τις δύο συνεισηγήτριες. Μέχρι τις 10 παρατέταρτο έχουμε χρόνο. Οπότε παρακαλώ πολύ, όχι πάνω από δύο λεπτά ο καθένας. Και Νάικελ. Ανώφελ. Θαυμάσια, θαυμάσια το είπατε το όνομά μου, που φαίνεται πως είναι κάπως δύσκολο για άλλους συμφωνώ με όσους, με τις ε, δύο κυρίες που μίλησαν πριν. Έχω ένα άλλο θέμα να θέσω υπόψη τη νομικής υπηρεσίας. Είπατε ότι η νομική βάση προβλέπει αφενός προστασία των θυμάτων και αφετέρου πρόληψη των εγκλημάτων. Τώρα, ανεξαρτήτως του τι είπαν οι προλαλήσασες, αυτή είναι η νομική βάση για την προσυπογραφή της σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ή της ισότητας. Βεβαίως και είναι η πρόληψη των εγκλημάτων σημαντική, αλλά το πιο σημαντικό από όλα δεν είναι να υπάρχει η βάση της ισότητας που να είναι ε, μια δυνατότητα διαβίωσης απαλλαγμένη από άσκηση βίας. Και από αυτό να προκύπτει ότι σαφέστατα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπέρ της ισότητας θέλω μια τοποθέτησή σας, γιατί νομίζω ότι ο περιορισμός σε προστασία θυμάτων και πρόληψη εγκλημάτων επιτυγχάνει ένα πράγμα. Βγάζει εκτός ότι πρόκειται για γυναίκες. Τα θύματα είναι γυναίκες και μάλιστα θύματα συστηματικής βίας. Δεν μιλούμε για οποιαδήποτε θύματα, ούτε για οποιαδήποτε άσκηση βίας. Μιλούμε για το μισό του ευρωπαϊκού πληθυσμού που υφίσταται συστηματική άσκηση βίας. Θα πρέπει λοιπόν πρώτα πρώτα να υπάρχει νομική βάση για την ισότητα. Ωραία, αν υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις για την νομική υπηρεσία θα τις θέσουμε όλες μαζί. Μάρλεν Μπιόρκ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τις δύο συνεισηγήτριες για τις παρεμβάσεις τους, με τις οποίες συμφωνώ. Να πω λίγα πράγματα από τη δική μου σκοπιά. Η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης είναι ένα πραγματικά φανταστικό νομοθέτημα και πολύ δύσκολο. Προέκυψε από πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις και την προσυπέραψαν όλες οι χώρες μέλη της Ένωσης και δέχονται ότι δηλαδή, αυτή η ε, άσκηση για έχει σχέση και με στερεότυπα ε, κυριαρχίας του άλλου φύλου. Αυτό το νομοθέτημα οφείλουμε να το υπερασπιστούμε και να είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό. Όλε οι χώρε μέλη το έχουν προσυπογράψει. Αλλά θέλουμε και να κυρωθεί. Και αυτό που είναι ανησυχητικό και κάπως ακούστηκε εδώ, ότι τώρα οργανώνεται αντίσταση. Δεν ειναι μεγάλε ομάδε, ομάδες, είναι οργανωμένε όμω. όμως. Είναι συντηρητικοί, είναι εθνικιστές, είναι σεξιστές, είναι αντι-LGBT κτλ. Και άλλε ομάδε του πληθυσμού. Και παίζουν με τα δικαιώματά μα. Κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο. Νομίζω λοιπόν, ναι, και Μπορούμε να συνεχίσουμε να συζητούμε για τα νομικά ζητήματα, τη νομική βάση κτλ. Αυτά όμως είναι βούτυρο στο ψωμί αυτών των ε, Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Ας βγούμε. Να διαμαρτυρηθούμε έξω από εκεί που, που συνεδριάζουν όλοι αυτοί. Εγώ είμαι εισηγήτρια στην Επιτροπή Γυναικών για ένα pilot project για την εφαρμογή των διατάξεων τη Σύμβαση Κωνσταντινούπολη υπέρ ε, μεταναστριών γυναικών. Και θα πρέπει όλε και όλοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και ξαναλέω να είμαστε υπερήφανοι για την Σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη. Και για μένα ω φεμινίστρια λέω ότι δεν μπορούμε να αντιτάξουμε δικαιώματα των μεν κατά δικαιωμάτων των δε. Λένε κάποιοι που αντιδρούν τώρα Α, να, η Σύμβαση Κωνσταντινούπολης δίνει δικαιώματα ε, σε διαφόρους ομοφιλοφίλους, ε, ε, καταστρέφει την παραδοσιακή οικογένεια. Δυστυχώς δεν τα κάνει αυτά η Σύμβαση Κωνσταντινούπολης, αυτό λέω εγώ. Όχι λοιπόν να βάλουμε, να μαλώνουν κειμένοι για τα δικαιώματα των δε και το αντίθετο. Οι δυνάμεις αυτές που κινητοποιούνται κατά τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης κινητοποιούνται και κατά των γυναικών και κατά των ομοφιλοφίλων. Είναι λοιπόν εχθρική απέναντι στις γυναίκες και εχθρική απέναντι στους ομοφιλοφίλους. Ο αγώνας λοιπόν πρέπει να είναι κοινό κατά των ανθρώπων αυτών. Έχοντας πει όλα αυτά, νομίζω ότι πρέπει να κινητοποιήσουμε και τους πολίτες στη συζήτηση αυτή. Κάτι το οποίο έχει άμεση σχέση με τις γυναίκες, με το δικαίωμα στο σώμα τους και οι γυναίκες είναι διατηρημένες να αγωνιστούν για να το στηρίξουν αυτά τα πράγματα. Ορίστε. Ε, κύριε Ρέιντκε, και εγώ συμφωνώ πρέπει να προχωρήσουμε από πολιτικής πλευράς έχει σχέση με τη λογοδοσία. Η βία εναντίον των γυναικών πολύ συχνά είναι αντικείμενο κηρυγμάτων ότι κάτι πρέπει να γίνει και να του τώρα έρχεται η στιγμή που μπορούμε κάτι να κάνουμε ε, και ταυτόχρονα ορισμένε κυβερνήσεις ε, κάνουν πίσω. Δύο ερωτήσεις προς την νομική υπηρεσία. Πρώτον, δεν είμαι νομικός. Ίσως θα προσπαθήσω να πω αυτό που νομίζω ότι είπατε με τα δικά μου λόγια. Εσείς κοιτάξατε όλη τη σύμβαση, ολιστικά δηλαδή, σφαιρικά, και αναζητήσατε νομική βάση ε, στις συνθήκες, στη συνθήκη. Ενώ το Συμβούλιο αυτό που έκανε είναι ότι κοίταξε συγκεκριμένες διατάξεις σύμβασης και για αυτές προσπάθησε να εντοπίσει προηγούμενα σε κοινοτικές οδηγίες ε, λέγοντας ότι στην πραγματικότητα έχουμε νομοθεσία ήδη. Ε, αν, κατάλαβα, αν σας κατάλαβα μάλιστα καλά, ε, ως αφορμή γι' αυτό το Συμβούλιο χρησιμοποίησε τη θέση, τη, την ιδιαίτερη κατάσταση της Ιρλανδίας και του Ενωμένου Βασιλείου. Δηλαδή αυτοί προσπάθησαν να μην ακολουθήσουν τη σφαιρική προσέγγιση επικαλούμενοι αυτή την, ε, αυτό το νομικό επιχείρημα το οποίο όμως δεν έχει βάσει συνθήκη. Δεύτερον, ε, όπως γνωρίζετε το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει και μια οδηγία για τη βία γυναικών και ένα από τα επιχειρήματά μας είναι ότι υπάρχει νομική βάση στις υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να αγωνιστεί υπέρ της ισότητας των δύο φύλων. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν και εγώ, αυτό θα μπορούσε να προστεθεί δίπλα στα άρθρα 82 και 84, δηλαδή σε μια ενδεχόμενη οδηγία για τη βία των γυναικών. Ο κ. Μωράης, ε, δεν έχουμε πολύ χρόνο, δύο μόνο ακόμα ομιλητές για να έχουμε και τις απαντήσεις. Κύριε Κοσλόφσκα, παρακαλώ. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις δύο συνσηγήτριες. Εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο δεν αμφιβάλαμε καθόλου για το ότι η Σύμβαση αποτελεί οδικό χάρτη για όλα τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση και η πρόοδος που έχει γίνει για να υπογραφεί η σύμβαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντική. Όλα τα κράτη-μέλη έχουν υπογράψει τη σύμβαση, οπότε θα ήταν παράξενο, τουλάχιστον, να γίνεται λόγος για έλψη προόδου ε, η σύμβαση αυτή έχει γίνει αναγνωριστή από τον ε, ΟΗΕ και από όλο τον κόσμο. Σε σχέση με άλλα έγγραφα, αυτή η σύμβαση συνδέει τις πολιτικές εναντίον της βίας με τις πολιτικές ισότητας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή τη σύμβαση. Πολλοί αγωνίζονται εναντίον αυτής της σύμβασης γιατί θεωρούν ότι η ισότητα ε, έρχεται σε σύγκρουση με την οικογένεια, ότι μια χειραφετημένη γυναίκα μπορεί να αμφισβητήσει το θεσμό της οικογένειας. Αυτό είναι λανθασμένο. Ποια οικογένεια λειτουργεί με βία, ποια οικογένεια λειτουργεί σωστά με βία, πώς είναι το να λέμε ότι αγωνιζόμενοι αντίον της βίας αμφισβητούμε ή υποσκάπτουμε την οικογένεια. Είναι πολύ σημαντική η αντίληψη που έχουμε για τη βία. 20% των Ευρωπαίων πολιτών θεωρεί ότι η βία, η ενδοοικογενειακή βία είναι κάτι εσωτερικό, ιδιωτικού χαρακτήρα. Θα πρέπει λοιπόν να να ε, ε, επιταχυνθεί επικύρωση από πλευράς των κρατών μελών προκειμένου να προχωρήσουμε στην πολιτική αντίον της βίας. Thank you very much. And finally, Mr. Jurek. πολύ, ο κ. Διουρέκ. Στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα βίας εναντίον των γυναικών. Ε, οι γάμοι η ε, υποχρεωτική γάμη, η έκθεση ε, σεξουαλικών πράξεων στο ίντερνετ που πολλές φορές αποτελεί βία εναντίον των γυναικών. Πριν από λίγο καιρό μάλιστα έγινε μια συζήτηση εδώ για τις ε, για τα αδικήματα τα οποία επέπεσαν ε, μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων στην ανθρωπιστική δράση. Ε, το... Ε, το σήμαση αυτή δεν τα περιλαμβάνει όλα αυτά ε, συγγνώμη, η νομοθεσία μας δεν τα περιλαμβάνει όλα αυτά, γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντική η σύμβαση. Θα ήθελα να πω ότι ε, δεν υπάρχει κανένα κράτος μέλος το οποίο να δέχεται στην νομοθεσία του ε, την ε, την ε, ύπαρξη ε, δυνατότητας ε, ενδοοικογενειακής βίας. Θα, θα ήταν παράξενο. Θα ήθελα να ρωτήσω αν πράγματι υπάρχει κάποια χώρα η οποία εισήλθε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με νομοθεσία η οποία να επιτρέπει την χρήση ενδοοικογενειακής βίας. Ε, στην, στην Πολωνία ε, υπάρχουν ε, πολλοί πολιτικοί, υπουργοί, ακόμα και πρωθυπουργό, που είναι εναντίον της επικύρωσης της σύμβασης, ότι θεωρούν ότι η σύμβαση είναι κοινωνικά επικίνδυνη. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από τους ε, από την νομική υπηρεσία να μας ε, ε, αναφέρει αν γνωρίζει κάτι τέτοιο και να μας πει ποιος είναι ο πραγματικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την επικύρωση αυτής της συμφωνίας. Έχετε το λόγο νομική υπηρεσία τώρα, δυστυχώ μόνο πέντε λεπτά για να απαντήσετε. Ε, thank you, Chair. I to be really very, very short ε, concerning the question on equality. νομικής υπηρεσίας. Για την ισότητα πολύ σύντομα. Πρόκειται για μικρό και επικουρικό μέρος της σύμβασης, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασίστηκε στα 82 και 84 της ΣΛΕ. Αντιλαμβανόμαστε την ανησυχία, αλλά δεν είναι από τα κυριαρχικά στοιχεία, τα κυρίαρχα μάλλον στοιχεία της ε, σύμβασης θα πρέπει να κάνει κανείς μια αντικειμενική ανάλυση του στόχου και του περιεχομένου της Σύμβασης Κωνσταντινούπολης και κάνοντας την ανάλυση αυτή η σωστή νομική βάση είναι το 82 για την προστασία των θυμάτων και ενδεχομένως το 84 για την πρόληψη των εγκλημάτων. Όσον αφορά το 77, το 77, νομίζω ότι είναι σωστή η ανάλυση του μέλου σας και το 78 για ε, το άσυλο είναι επικουρικού χαρακτήρα πάλι στα πλαίσια της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Θεωρούμε λοιπόν ότι δεν είναι κατάλληλα να ληφθούν υπόψη ως νομικές βάσεις για να θα δικαιολογούσαν έτσι και την διάσπαση. Σχετικά με το έγγραφο που ζητήσατε, έχουμε διαβιβάσει τη νομική ε, γνωμοδότηση. Ίσως υπάρχουν και άλλα έγγραφα τα οποία είναι και δημόσια έγγραφα ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Συμβουλίου σχετικά με την ίδια τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης που είναι βεβαίως στη διάθεσή σας και εμείς είμαστε στη διάθεσή σας να τα δώσουμε. Τέλος, για την ε, οικιακή βία. Η νομική υπηρεσία προπενταετίας, ίσως και λιγότερο, είχε εκδώσει γνωμοδότηση για την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό. Είναι σαφές ότι η οικιακή, μάλλον ο αγώνας κατά της οικιακής βίας είναι καταρχήν αρμοδιότητα των χωρών μελών και όχι της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας παραπέμπω σε αυτή τη νομική γνωμοδότηση την οποία συντάξαμε για λογαριασμό της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών ε, τότε. Ε, αυτά είναι όλα, δεν ξέρω αν ο αδερφός μου, ο οποίος όμως μεύει αποφατικά, θέλει να προσθέσει κάτι. Οτιδήποτε άλλη πληροφορία στη θέση σας. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος Μωράς. Δεν έχουμε πια πολύ χρόνο. Πολύ σαφώς πάντως από την πλευρά της Επιτροπής Θεμελιωδών Ελευθεριών παρακολουθούμε προσεκτικά τις τοποθετήσεις και των δύο συνεισηγητριών και τις διευκρινήσεις για την νομική βάση. Τίποτε στη νομική γνωμοδότηση δεν υπάρχει που να λέει ότι προχωρούμε με τον κώδικα διοντολογίας για την Λίμπε λοιπόν είναι σαφή τα πράγματα αυτά και όπως είπε η κυρία Μπιόρκ θέλουμε να περιληφθούν και άλλα θέματα, ισότητα κλπ. Ό,τι υπάρχει μέσα πρέπει να προχωρήσει. Δεν χρειαζόμαστε ε, μακροσκελείς νομικές νομοδοτήσεις τις οποίες περιέμεναμε και το καιρό και μετά να τις έχουμε και να μην προχωρήσουμε. Υπάρχει σαφής πλειοψηφία για να προχωρήσουμε. Θα γράψουμε λοιπόν πρώτα στη Βουλγαρική Προεδρία να θέσουμε ερωτήσεις και να πιέσουμε να προχωρήσουν αυτά που ζητούν οι δύο συνεισηγητρίες. Δεύτερον, για τον κώδικο δεοντολογίας και το σχέδιο κύρωσης. Να δηλώσουμε ότι αυτή είναι η επιθυμία μας και οποιαδήποτε πρόσθετα μέτρα οφείλουν να ληφθούν. Θα ρωτήσω τις συνεισχύτριες αν έχετε άλλες ιδέες να τις προωθήσουμε, διότι τώρα βέβαια έχουμε κάποια πίεση χρόνου. Πλησιάζουμε άλλωστε και στο τέλο τη ε, τρέχουσα Προεδρία και στην αρχή τη Επόμενη. Είναι σαφέ για την Επιτροπή μα την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, ότι δεν υπάρχει τίποτα στην νομική γνωμοδότηση που να αποτρέπει από το να ε, συνεχίσουμε αυτά στη νομική βάση που ε, αναφέρατε. Ορίστε εσείς τώρα. Ευχαριστώ τους εκπροσώπους νομικής υπηρεσίας. Πρώτον, λέει η κυρία Μπλίνκεβιτσιούτε για την παρουσίαση γνωμοδότησής τους. Ευχαριστώ και τις δύο συνεισηγήτριες που ε, παρενέβησαν, καθώς και όλα τα μέλη. Υπενθυμίζω, για λογαριασμό της Επιτροπής Δικαιωμάτων Γυναικών, ότι στις 10 η ώρα έχουμε συνάντηση των συντονιστριών και μετά αρχίζει η συνεδρίασή μας. Ευχαριστώ πολύ, Κλοντ, για την φιλοξενία.